στη σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπείων, ο αντίστοιχο κατάλογο θα προσαρτηθεί στα πρακτικά τη σημερινή συνεδρία. Εάν στην έγκριση των πρακτικών δεν υπάρξει καμία αντίρρηση, τότε αυτέ οι τροποποιήσει θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί. Βάσει του άρθρου